Sí, buenos días a todos. Eh, vamos a empezar la, la reunión de la Καλημέρα σας, λέει πρόεδρος. Πρώτα, πρώτα, θα συζητήσουμε το 10ο σημείο της διατάξεως. Για να δούμε τα σχετικά με την διμερή αλληλευτική συμφωνία ΕΕ και Πρασινού Ακροτηρίου. Όπω γνωρίζετε, εισηγητής ο κύριο Γκάλα. Οπότε, ο και αυτό μάλλον, στον οποίο θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο. Α, α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρώτα πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο η οποία να μα κάνει την εισήγηση τη σχετική με αυτό το σημείο. bueno, usted tiene la palabra. Merci, Madame la Présidente. Euh, Έχουμε αυτό το καινούργιο πρωτόκολλο με την εν λόγω χώρα, το πράσινο ακροτήριο, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει μονογραφηθεί, έχει υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 10. Θα είναι τριετής η διάρκεια του και θα τεθεί σε ισχύ ε, από την ημερομηνία που εκπνέει ισχύουσα συμφωνία, δηλαδή πρώτης ένα του τώρα αυτό που ενδιαφέρει είναι εκείνη η ρήτρα μέσω της οποίας μπορούμε να αναστείλουμε την συμμετοχή της χώρας και σε περίπτωση που τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αρχές δεν σέβονται, αναστέλλεται συμφωνία ως προς την εν χώρα. Πέραν αυτών τώρα. Εδώ έχουμε ένα χτένισμα των δυνατοτήτων αλίας συνεχίζουμε να έχουμε 5.000 ε, τόνους και έχουμε être pour répondre de manière plus réaliste aux besoins euh, de la flotte. Και επομένως με αυτές τις ε, τράτες επιφανείας ε, μπορούμε να κινηθούμε ως ευρωπαϊκός αληθικός τόλος. Αυξήθηκε επομένως η δυνατότητα που προέβλεπε η παλιότερη συμφωνία και αυτό διότι αυξήσαμε και τα ποσά τα οποία αφορούν αυτόν τον κλάδο. Και σύμφωνα με όσο προβλέπονται τώρα έχουμε 60.000 ε, ε, ευρώ και τα 60 γίνανε στη συνέχεια 110.000 τα οποία χρειάζεται η χώρα και έπρεπε επομένω να γίνει αυτή η αύξηση της δικής μας συμβολής και έτσι να προσπαθήσουμε να συμμετάσχουμε πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την αλληλεία στο πράσινο κροτήριο. Ένα άλλο στοιχείο τώρα που αφορά αυτό το νέο πρωτόκολλο. Όσον αφορά τώρα το ποιοι προσλαμβάνονται στα ελληνικά, θα πρέπει να είναι οι θαγενείς της χώρας. Επομένως δεν αυξάνεται ο αριθμός των σχετικών αυτών. Πριν ήταν ναύτες ΑΚΕ, τώρα όμως θα είναι ναύτες της ναυτική τέλο πάντων της χώρας. Επίσης η χώρα δέχθηκε να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε κάποια σκάφη ανοιχτής θαλάσσης. Επίσης προβλέπεται ένα πρωτόκολλο VMS για εποπτεία μέσω δορυφόρου. Επομένως τώρα τα πράγματα θα ρυθμίζονται με πολύ πιο ενδελεχή τρόπο, γιατί όσον αφορά την ε, εποπτεία είχε πρόβλημα αυτή η χώρα. Και τώρα θα ισχύσει αυτή η ρύθμιση ε, μόλις με την ε, δική μας υποστήριξη μπορούν να είναι λειτουργικά τα σκάφη τους. Επομένως αυτή του είδους η χρήση δορυφόρου θα ισχύσει για όλα τα σκάφη τα οποία αλλιεύουν ε, στα χωρικά έδατα της χώρας αυτής. Όσον αφορά τώρα τους ε, πλειοκτήτες έχουμε μια ελαφρά αύξηση όσον αφορά την ε, τιμή της αδείας. Τώρα καλύπτονται ακόμα περισσότεροι τόνοι που καλύπτει σχετική άδεια, σχετική έγκριση. Θα υποβάλουμε αυτό το σχέδιο κανονισμού στο Συμβούλιο. Ε, θα συζητηθεί και θα εγκριθεί, ελπίζουμε, στις 9 Ιουνίου. Αυτό δεν είναι σίγουρο ενδεικτικά μας είπε ότι αυτό θα γίνει στο Συμβούλιο και θα υπάρξει αυτή η υπογραφή και με τους εκπροσωπητές της χώρας. Ε, αυτό δεν θα πάρει πολύ χρόνο γιατί εκπροσωπούνται στις Βρυξέλλες ή του Πρασίνου Ακροτηρίου, οπότε και θα προχωρήσουμε σε αυτή την υπογραφή της συμφωνίας που προβλέπεται να κάνει το Συμβούλιο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. θέλετε eh, τώρα το λόγο ή στο eh, eh, Ό,τι θέλετε, και τώρα και μετά. Ωραία, ah, um, Ευχαριστώ την Επιτροπή για την σύντομη σύνοψη που έκανε. Είναι προφανές ότι είναι πολύ σημαντικό να μην καθυστερήσουμε την έγκριση αυτής της ανακοίνωσης ε, στο Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η υπάρχουσα συμφωνία εκπνέει την 1η Σεπτεμβρίου και πρόκειται για μια συμφωνία που είναι σημαντική τόσο για το πράσινο ακροτήριο όσο και για τους, τον ευρωπαϊκό στόλο. Ε, πολλές συμφωνίες κατά κάποιο τρόπο επεκτείνονται και το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση, αλλά πρέπει να πω ότι χαίρομαι που έχουν περιληφθεί κάποιες ε, τροπολογίες, διότι έχουν ληφθεί υπόψη συστάσεις όχι άλλων επιτροπών αυτού του Κοινοβουλίου, αλλά της Επιτροπής αλληλία και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν μπορεί να ανασταλεί η καταβολή αν παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή δημοκρατικές διαδικασίες. Χαίρομαι επίσης για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς το σύστημα επιτήρησης των σκαφών και ε, το σύστημα αδειοδότησης και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί. Ενώ το συνολικό ύψος φτάνει στις 5.000. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν από την Κομισιόν στη φάση αυτή αν η ζήτηση ε, μεταξύ των ε, παραγαδιών επιφανίας και των ε, άλλων θυναλιευτικών. Η ζήτηση είναι μεγάλη. Πρέπει να παραμείνουμε αυστηρος στο όριο των 5.000 ή μπορεί να υπάρξει κάποια ευελιξία. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Και πιστεύω ότι θα είναι εποφελής τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το, και το Πράσινο Ακροτήριο. Επίσης είναι σημαντικό το ότι οι αλλοίς από το Πράσινο Ακροτήριο μπορούν να συμμετάσχουν. Ε, λέτε μπορεί, μέι, ε, μήπως είναι μάστε ότι πρέπει. Δηλαδή και άλλοι συμμετείχαν προηγουμένως πριν από αυτή τη συμφωνία. Και επίσης θα έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ε, βοηθητικών σκαφών που μέσω της συμφωνίας που υπογράφεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκύψει κάποιο όφελος και για τα βοηθητικά σκάφη. Συνολικά λοιπόν η όλη συμφωνία δείχνει απολύτως αποδεκτή και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκάλαγκερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι για το θέμα της συμπερίληψης του VMS και την ρήτρα περί τήρησης των σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, με ανησυχεί το θέμα της αξιολόγησης και το πώς αυτή εφαρμόζεται. Μία από... Ένας από τους λόγους της διατήρησης των FPAs είναι να βοηθήσουμε τις χώρες εταίρους σε θέματα ελέγχου και εποπτείας, επιτήρησης. Και διαπιστώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Αλληλείας στο Πράσινο Ακροτήριο δεν διαθέτει καθόλου μέσα ελέγχου και επιτήρησης και όλες αυτές οι αρμοδιότητες έχουν δοθεί στο λιμενικό ε, και στο στρατό που και επίσης δεν έχουν δυνατότητες. Υπάρχουν δηλαδή δυσκολίες στο να διατηρηθεί η, ε, στο να υπάρξει επαρκής έλεγχος ε, και οι περιπολίες που γίνονται από το λιμενικό στα παράκτια δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα και η επικοινωνία η επικοινωνία δε μεταξύ λιμενικού και αρμοδίων αρχών δεν είναι ε, επίσημη, τυποποιημένη. Συνεπώς δεν είναι λειτουργικός αυτός ο έλεγχος. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ένας άλλος παράγων, πολύ ανησυχητικός, που προκύπτει από την αξιολόγηση, είναι η ρήτρα αποκλειστικότητας. Στο πράσινο ακροτήριο έχουμε μία όμορη περιοχή με χίλια σκάφη και τρεις χιλιάδες αλληλείς και επιπλέον υπάρχουν δύο ισπανικά γρηγροί. Ε, οκτώ δέκα χιλιάδων τόνων ε, παραγωγής ετησίως. Κατά πάσα βιδανότητα, όχι στα ύδατα του πράσινου ακροατηρίου, αλλά πηγαίνουν στην ακτή ε, του ελεφαντοστού. Ε, και εκεί έχουμε ρήτρα αποκλειστικότητας. Και εδώ αναφέρεται ότι είναι ισπανικά σκάφη. Θα μπορούσε λοιπόν να διευκρινίσει η Κομισιόν πώς αυτά τα σκάφη λειτουργούν σε αυτά τα ύδατα, αν υπάρχει ρήτρα αποκλειστικότητας τότε όλα τα ευρωπαϊκά σκάφη θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τη συμφωνία ακόμα και με σημαίες άλλων χωρών εξ όσων εγώ αντιλαμβάνομαι και θέλω μια διευκρίνηση. Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα το οποίο επί συζητήσαμε είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, αντιμετωπίσει την αλία π λάμδα αλφα παγκοσμίω. Ωστόσο, η αλλιεύσεις, η ποσότητα των αλλιευμάτων δεν είναι επαρκή. Ψάρια εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται η επεξεργασία στο πράσινο κροτήριο και μετά επανεξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και οι αρχικοί έλεγχοι δεν γίνονται επαρκώς και υπάρχει ο κίνδυνος ε, προμήθειας αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μη εγκεκριμένε πηγές, δηλαδή πηγέ πι Πώς λοιπόν η Κομισιόν δεν προσέφερε επαρκή υποστήριξη στο πράσινο ακροτήριο για να ξεκαθαρίσει τις πηγές των ηχθείων που, των οποίων η επεξεργασία γίνεται πάνω στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό προκύπτει από την αξιολόγηση. Επιπλέον, δεν έχουν μπει παρατηρητέ στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είπατε, όχι δεν είπατε, είπατε για το πλήρωμα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θα υπάρχουν παρατηρητές πάνω στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην προηγούμενη συμφωνία δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στα VMS, αυτό είναι πολύ σημαντικό. αυτό ε, έλειπε και ήταν εξοργιστικό που δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος των σκαφών. Τώρα, η ε, συντήρηση, γιατί ένα στόχος είναι και αυτή ένα στόχος είναι η βιώσιμη αηφόρος αλληλεία. Αν ε, κοιτάξει κανείς τα, το τι αλλιεύεται, Ε, είναι ok για την Παλαμίδα, αλλά ως προς τον τόνο η αντικατάσταση της ε, προηγούμενης απαγόρευσης ε, για τα είδη αυτά είναι λιγότερο αποτελεσματική για τα νεογνά. Συνεπώς πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα για τα ε, ηχθίδια, για τα νεογνά ψάρια του τόνου Big Eye. Και Έχουμε επίσης και κάποιες... Ε, And uh, as bycatch. Έχουμε κάποιους καρχαρίες που είναι κάποια είδη καρχαριών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ως προς τις απορρίψεις τώρα, υπολογίζεται το 22% απορρίπρεται, δηλαδή ε, σκουμπριά, ε, παλαμίδες, μακρόπτερη τόνη κλπ. 22% λοιπόν. Τι προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μείωση των αλλιευμάτων που απορρίπτονται. Τώρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με την τομεακή υποστήριξη που χορηγείται επιπλέον της άλλης αρρωγής που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει επαρκή συντονισμός μεταξύ ευρωπαϊκής ε, στήριξης και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και των άλλων μέσων στήριξης. Και οι σύμβουλοι θα λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα περιφερειακό συντονιστικό έργο και όχι ένα εθνικό. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστούμε την Επιτροπή, ευχαριστούμε και τον κύριο Συγητή. Εγώ θα σα πω ότι για αυτή την έκθεση αξιολόγηση που όπως και η κυρία Λόβιν και εγώ με μεγάλη προσοχή την μελέτησα, είδα στα συμπεράσματα ότι είναι πάρα πολύ θετική η κατάληξη της έκθεσης αυτής, ακριβώς όσον αφορά το τι θα κάνουμε σε κάθε περιφέρεια στην Ανατολική Αφρική όσον αφορά τον τόνο. Επίσης, θετικά αξιολογούνται οι δυνατότητες αλλίες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες εις τις ανάγκες. Όσον αφορά το με, τον μέσο όρο απορρόφησης, το σχετικό ποσοστό, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε αύξηση της ζήτησης, κυρίως όσον αφορά την παράκτεια αλεία. Είχαμε επίσης και αύξηση της ζήτησης στον Ινδικό, είχαμε επίσης και πλήγματα από την αύξηση της πειρατείας και έτσι τώρα αυξάνονται οι ανάγκες όσον αφορά την Ανατολική Αφρική. Έχουμε από Γαλλία, Ισπανία, ε, Γαλλία, αληφτικά, τα οποία εκεί αναπτύσσουν δραστηριότητα. Έχουμε από 25 σε 28 αυτή την αύξηση όσον αφορά την παρακτή αλληλεία. Και έτσι όσον αφορά τις τράτες έχουμε μία προσαρμογή προς τα κάτω. Και επίση είπαμε πάμε στο 84% όσον αφορά το, το κόστος των εγκρίσεων. Τώρα, ακούσαμε τι είπε η κυρία Λόβιν για τα σκάφη που λέγονται ισπανικά, αλλά έχουν σημαία πρασίνου ακροτηρίου παρά το ότι χρηματοδοτούνται από Ισπανούς αυτές οι δραστηριότητες. Πάντως, να σας τα εξηγήσω αν θέλετε, αλλά δεν πάνε καν εκεί. Και πρόκειται για σκάφη τα οποία φέρουν σημαία του πρασίνου ακροτηρίου. Επίσης, Όσον αφορά αυτή την επιχείρηση, είναι ισπανική. Και ακριβώς για να τηρηθούν οι διατάξεις σχετικές με την προέλευση, εισάγονται πρώτες ύλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς αυτή η εταιρεία συμμορφούμενη με τις διατάξεις για την προέλευση. Ανοίγει στην ICAT το πράσινο ακροτήριο. Και βέβαια θα πρέπει και εκείνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφώνουν με σχετικέ διατάξει. Επομένω εδώ δεν έχουμε θέμα διατήρηση των πόρων και συντρέχουν, ξαναλέω, οι διατάξει τη ΕΚΑΤ. Για πέστε μας για τους ναυτικούς. Για πέστε μας, ε, εκπρόσωπε της Επιτροπής, Ακριβώς επειδή είχαμε την ε, εστίασή μας στην, στις, στις περιφερειακές και είχαμε και κάποια μεταναστευτικά είδη, είχαμε πει ότι έχουμε κάποια ελευτικά τα οποία έχουν άδεια να αλλιεύουν σε όλη τη ζώνη. Να μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις των ψαριών και ακριβώς γι' αυτό και δυνάμει των σχετικών συμφωνιών και είχαμε αύξηση του πόσοι θα συμμετέχουν ναυτικοί από κάθε ε, από κάθε χώρα, δηλαδή από ΕΟΚ, από ΑΚΕ λοιπά Τώρα είπαμε ότι άλλαξε και πάλι. Και είπαμε ότι θα πρέπει να προέρχονται από το πράσινο ακροτήριο και να υπάρχουν σχετικές άδειε τώρα προβλέπεται. δηλαδή τώρα ξαναγυρίζουμε στο παλιό καθεστώς. Δεν βλέπω να υπάρχει εδώ ικανοποιητική αιτιολόγηση του γιατί γυρίσαμε στην παλιά ρύθμιση. Για πέστε μας. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει γιατί τώρα δεν ισχύει το παλαιότερο ευέλικτο καθεστώς το οποίο κάλυπτε ακριβώς τις ανάγκες των σκαφών που εκεί ανέπτυσαν αλληλευτική δραστηριότητα. Μισό λεπτό, δεν ξέρω το όνομά σας, δεν ξέρω αν θα το προφέρω ε, σωστά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν ανοίγεται μερικά ονόματα που είναι δύσκολα να τα προφέρω. Θα ήθελα ωστόσο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν. Καταρχήν όσον αφορά το υφό, όσον αφορά τους τόνους αναφοράς και το περιέχον τόνων. Στο σύνολο έχουμε βεβαίω πολύ λιγότερα πλοία, σκάφη σε αυτό το νέο πρωτόκολλο, πρωτόκολλο συγγνώμη, και το θέμα το οποίο τίθεται είναι τα επόμενα, στα προηγούμενα 4,5 χρόνια που δίρκεσε το πρωτόκολλο αυτό, είχαμε στο σύνολο είχαμε αυτά τα περίπου τον αριθμό, αυτό τον αριθμό των πλοίων τα οποία αναφέρθηκαν και το ανώτατο όριο αλίευσης ήταν 3.400 τόνοι. Σε αυτά προσθέσαμε βεβαίω σε αυτό προσθέσαμε και άλλα ποσά, διότι και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε ο, οι τόνοι αναφορά να μειωθούν για να καλύπτονται έτσι τα πράγματα όσον αφορά το πρωτόκολλο. Και έτσι φτάσαμε τους 5.000 τόνους. Τώρα, όσον αφορά την υποχρέωση που υπήρξε, δεδομένου ότι είναι μία η, υποχρέωση να υπάρξει μπαρκάρισμα αλλιέων που ήταν από το πράσινο κροτήριο, ξέρετε πόσα χώρα αυτή δεν θέλησε να υποχωρήσει. Για αυτούς υπήρξα ζωτική σημασίας και να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να υπάρχουν μέσα εκεί ε, αλληλείς οι οποίοι είναι από τη χώρα αυτή, από το, από το πράσινο ακροτήριο. Και βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιβάλλουμε για κάθε συμφωνία. Δεν μπορούμε βεβαίω να επιβάλλουμε το ανώτατο όριο αλλιέων οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσα στο πλοίο. Τα μπαρκάρουν δηλαδή. Πρέπει να είναι ένα περιορισμένο αριθμό, ο οποίο θα εφαρμόσει σε όλο το στόλο και θα είναι για 114 σκάφη. Υπάρχει υποχρέωση 13 αλλιέων από τη χώρα αυτή το Πρασοκρατήριο. ή αυτοί μπαρκάρουν και υπάρχουν. Και νομίζω δεν είναι μόνο 13 όπως είναι η υποχρέωση, η γραφτή υποχρέωση, αλλά περισσότεροι μάλλον. Άρα ήταν ένα θέμα για το οποίο το πράσινο ακροτήριο ήταν διατεθειμένο να διαπραγματευτεί. Υπάρχει βέβαια κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να δεθεί και το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Φρονώ όμως ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε μια συνεργασία, σε μια γνήσια συνεργασία με αυτή τη χώρα, ούτως ώστε για να υπάρξουν μαζί τα, μια κοινή επίβλεψη και έλεγχος οι δράσει της περιοχής. Υπάρχει μια επιτροπή η τοπική για τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, η οποία εδράζεται στο Ντακάρ και η οποία βεβαίω είναι πιο απαιτητική και δέχεται την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Υποστήριξης και προς στιγμή είναι μια ομίγυρης διαλόγου, συζητήσεων κλπ. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε υπόψη μας τα δεδομένα εκείνα τα οποία σε μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, αλλά ακόμη τα πράγματα δεν έχουν φτάσει αυτή και σε αυτό το σημείο και οι χώρε αυτέ δεν είναι διατηρημένε να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Τώρα, όσον αφορά το πράσινο ακροτήριο, θα πρέπει να πούμε ότι είναι το πρόβλημα. Είναι μια μικρή χώρα, όπως ξέρετε, που έχουν τεράστιες ανάγκες, δεν έχουν τα μέσα τα οικονομικά, δεν έχει η Γενική Διεύθυνση αλλήλεια δεν έχει δύο σπόρους και βασίζεται στην ακτοφυλακή και μόνο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δημιουργούν ένα μεμοράντουμ, ένα υπόμνημα όσον αφορά την ακτοφυλακή και Είχαμε προβλέψει βεβαίω να, να δοθούν κεφάλαιο επιδοτήσει σε αυτό το θέμα. Τώρα κάνουμε κάτι άλλο. Κάνουμε ένα βήμα παρετέρω, πιο πάνω, για να υπάρξει ένα υπόμνημα memorandum με τους πρασινοακτήτες και θα πρέπει να ζητήσουμε ούτως ώστε η πράσινο ακτή και η γενική της διεύθυνση να έχει τη δική τη ομάδα ελέγχου και αυτοφυλακή. Θα πρέπει αυτοί να το έχουν. Βέβαια δεν θα γίνει αυτό εντάχει. Πλην όμω, εάν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή για να γίνει αυτή η συνεργασία, να γίνει πιο συστηματική, να υπάρχουν κανονισμοί, τότε ενδεχομένω θα έχουμε κάτι καλύτερο από ό,τι σήμερα. Ελπίζοντα βεβαίω να γίνει κάτι τέτοιο, καθώ επίση και ένα σύστημα το οποίο θα είναι μια δορυφορική παρακολούθηση, την οποία εμεί την έχουμε θέσει σε λειτουργία και παρακολουθούμε τα πράγματα. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα έχουμε πρόοδο στο μέλλον στα θέματα αυτά. Ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται είναι το θέμα των παρατηρητών. Ξέρετε ότι το πράσινο ακροτήριο δεν υπήρξε σε θέση να βάλει παρατηρητές επί των σκαφών, των πλοίων και ζητήσαμε εμείς, είπαμε λοιπόν εμείς, δεν μπορούμε να δράσουμε στη θέση της χώρας αυτής. Κάνουμε λοιπόν ένα νέο πρωτόκολλο το οποίο θα προβλέπει ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν παρατηρητές και όπου εμείς συμβάλαμε πάρα πολύ, όπου βάλαμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε ακόμη περισσότερε από αυτούς που χρειάζονται, πράγμα το οποίο θα μα επιτρέψει να έχουμε ένα μάτι θα λέγαμε σε αυτά τα πράγματα, στο τι συμβαίνει και μεταξύ εκείνων των μέτρων τα οποία έχουμε θέσει είναι να έχουμε, ιδιαίτερα επιμένουμε στο να έχουμε τον παρατηρητή πάνω στο σκάφος, να, βλέπουμε, να παρακολουθούμε εκ του τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά στις, ε, παράπλευρες, παράπλευρη αλίευση παρεμπίπτοντα αλλιεύματα πιστεύω πως η ταχύτητα της, α, της αλίευσης είναι τέτοια, είναι πραγματικά αλήθεια ότι υπάρχουν ορισμένα είδη τα οποία έχουν υπεραλλιευτεί. Εν πάση περιπτώσει τα δικά μας αλλιεύματα είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση με τα ποσά της ερήψης που γίνεται όσον αφορά την ηλικία των ε, αλληλευμάτων διορθώται κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν θα πρέπει, κατά πόσο θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ινστιτούτα της αλήψης αυτής της χώρας, καθώς επίσης και με τους επιστήμονες που εργάζονται στην, στο πράσινο ακροτήρι. Τώρα, όσον αφορά τα ισπανικά πλοία, σκάφη. Πρόεδρε, όντως όντως, συμφωνούμε μαζί σας ότι τα πλοία αυτά έχουν σημαία πρασίνου ακροτηρίου. Είναι μια δραστηριότητα της χώρας αυτής. Δεν είναι ισπανικά. Δεν είναι λοιπόν της δικής μας αρμοδιότητας, δεν είναι της δικής μας κάλυψης του χώρου αυτού. Και βεβαίω αυτό το, δεν άπτε του δικού μας κανονισμού, εφόσον δεν είναι διποδική μας σημαία. Τέλος, όσον αφορά την μεταποίηση των πλοίων αυτών και την εκφόρτωση και τη μεταποίηση των πλοίων αυτών αυτών των ψαριών, των ψαριβάτων, τα δεν αφορούν τον τόνο αυτά, αυτές οι μικροβιομηχανίες που υπάρχουν εκεί. Δεν μεταποιούν τον τόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να ξεφορτώσουμε εμείς τα δικά μας ψάρια για να τροφοδοτήσουμε αυτή τη βιομηχανία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους ότι παρά τα κίνητρα τα οποία έδεσε η χώρα αυτή, το πράσινο κροτήριο, εμείς δεν κάνουμε εκφόρτωση αυτών των ψαρών, καθότι δεν υπάρχουν αγοραστές στη χώρα αυτή. Φρονώ λοιπόν πώς έχω απαντήσει τα ε, στα ερωτήματα που ετέθησαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάλαγερ, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Άκουσα προσεκτικά τα όσα ελέγχθησαν, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η καθυστέρηση ως προς την ε, χρησιμοποίηση των παρατηρητών. Μέρος της δουλειάς των παρατηρητών <coughs> είναι ακριβώς να παρακολουθήσουν την, ε, τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα και τις ε, απορρίψεις. Και δέχομαι απολύτως ότι σε μια ιδανική κατάσταση αν οι τόνοι έρχονταν στην ακτή και η επεξεργασία γινόταν εκεί, ε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ωστόσο δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για την επεξεργασία πελαγικών ηχθείων και αυτό που απαιτείται είναι τεράστια επένδυση και δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Και ούτε διαθέτουν και τον εξοπλισμό το δορυφορικό για την παρακολούθηση που είναι απολύτως απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση. Και υπάρχει όμως ένα μνημόνιο συναντήληψης με το πράσινο ακροτήριο και η Κομισιόν θα συγκροτήσει, ε, θα συντάξει φαίνεται ότι θα το ένα νέο μνημόνιο συναντήληψης. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ε, θα ήθελα βέβαια να μάθω, ε, αλλά αυτό αφορά μία ιδιωτική συμφωνία. Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς έχει γίνει με τους Ιάπωνες που διαθέτουν παραγάδια επιφανίας και που ψαρεύουν στις θάλασσες αυτές και να κάνουμε και μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Ιαπώνων και ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει προσβλέπω στην θέση σε ισχύ του νέου πρωτόκολλου τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, διότι αν δεν υπάρξει πρωτόκολλο ή συμφωνία θα υπάρχει ένα κενό, διότι το ισχύον πρωτόκολλο εκπνέει όπως σας είπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε απλώς πρέπει να σας αναφέρω ότι στις 15 Ιουνίου θα εξεταστεί το σχέδιο κειμένου, 12 Ιουλίου θα γίνει η ψήφιση και καταρχήν πρόκειται να περάσει από την πρώτη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώσαμε τώρα το σημείο υπαριθμών 10. Πάμε στο επόμενο, το οποίο αφορά τη Σύμβαση Διατήρηση και Διαχείριση Ελεκτικών Πόρων Ανοιχτής Θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. η ομιλούσα είναι η συγκίτρια. Θα μας παρουσιάσει αυτή την ε, σύμβαση ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Πραγματικά εξετάζουμε σε τη στιγμή με τη σύμβαση ως αρφα τη διατήρηση και την τους πόρους και τις υδροκαλλιέργειες που βρίσκονται στο, στα ανοιχτά του νοτίου ε, ειρηνικού. Κάθε πώ θα γίνει η διατήρηση. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπήρξε μια ιστορικό όσον αφορά τη διαπραγμάτευση θέση του πρωτοκόλου που ξεκίνησε το 2006 η Αυστραλία η Χιλή, η Κίνα. Ε, ξεκίνησα μια προσπάθεια ό, όσον αφορά αυτά τα είδη τα οποία βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα του Νοτιού Ειρηνικού Ωκεανού ιδιαίτερα εκείνα τα είδη τα οποία καλύπτονται αυτά τα, από την σύμβαση συμφωνία αυτή, το σύμφωνο αυτό μάλλον καλύτερα. Σκοπός αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, ότι βοήθησε πάρα πολύ ο μα σε αυτή την υπόθεση, όπως σας είχα πει από το 2006, για αυτή τη διεθνή διαπραγμάτευση και την συμφωνία, η οποία περατώθηκε το Νοέμβριο του 2009. Αυτή υπογράψαμε, προσυπογράψαμε λοιπόν αυτή τη σύμβαση τον Ιούλιο του 10. Προφανώς αυτή τη στιγμή είναι ένα σύγχρονο εργαλείο γιατί υπάρχουν ξέρετε πάρει εξελίξεις οι οποίες έχουν γίνει στον τομέα της αλληλείας όπως εκμεταλλευτήκαμε τις συμφωνίες που έχουν γίνει όσον αφορά την τον κεντρικό ελληνικό ωκεανό, όλη την εμπειρία την οποία έχουν, καθώς επίσης και τη διαχείριση όλων αυτών των αλλιευμάτων που έχουν αυτές. Για να αναφέρω ορισμένα από αυτά, το οικοσύστημα, την προληπτική ε, προσπάθεια που γίνεται, άρθρο 3, όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, η, προ, η τα στάνταρτα τα οποία πρέπει να υπάρχουν για αυτό το χώρο, τον τρόπο για την συντήρηση και διατήρηση ολυμένων αλλιευμάτων, καθώς επίσης και τη διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθείτε, το, το οποίο κατά την άποψη της Κομισιόν είναι ένα από τα καλύτερα επιτεύγματα αυτή της προσπάθειας η οποία έχει γίνει, καθώς επίσης και του συμφώνου και παίξαμε ένα αποφασιστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση αυτή εμείς σαν Κομισιόν. Αυτή η απόφαση λοιπόν είναι μια διαδικασία απόφαση η οποία ξεκίνησε από συνένεση, αλλά ωστόσο υπήρξε υπήρξε μια, ένας αυτοσχεδιασμός όσον αφορά την, ψηφο, την ψηφοφορία. Υπήρξε μια διαδικασία η οποία ήταν, που δεν έπρεπε να πάμε περι, περαιτέρω από αυτή και υπήρξαν απορρίψεις πραγμάτων. Υπήρχαν αντιρρήσεις οι οποίες θα πρέπει να λειτουργήσουν υπόψη και εάν Κάποιο αντιτίθεται σε αυτά τα μέτρα τα οποία δεν θέλει να δεχθεί θα πρέπει να λαμβάνει άλλα μέτρα για να μην υπάρξουν διακρίσεις. Έτσι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα που διασφαλίζει κατά αυτόν τον τρόπο την τήρηση τη συμφωνία. Υπάρχουν τα θέματα της ε, αναγνώρισης, της διαφάνεια όσον αφορά τα Υπάρχουν ε, άρθρα τα οποία έχουν αρκετή ελαστικότητα όσον αφορά την εφαρμογή τους, καθώς επίσης παρατηρητήρια, ομάδες παρατήρησης, αυτό που προσπαθώ να πω, υπάρχουν ε, πολλά πολλά στοιχεία τα οποία, στα οποία κανονικά στις παλιές συμβάσεις δεν υπήρχαν στη δευτερεύουσα τουλάχιστον ε, και την παράγωγη θα λέγαμε στα ελληνικά νομοθεσία εισάγονται. Αντιθέτως αυτή τη στιγμή τα βρίσκουμε στο βασικό κείμενο της εμφανίσης. Υπάρχει ένα πρόγραμμα παρατήρησης όπως σας είπα, ένα πρόγραμμα ελέγχου και όλα αυτά βρίσκονται μέσα τη συμφωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτή την υπόθεση. Η ΕΕ λοιπόν έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα και συμφέροντα στο νότιο ειρηνικό. Έχουμε λοιπόν σύμφωνα με τη Συμφωνία της Νέας Υόρκης να συνεργαζόμεθα με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τους αλληλευτικούς σπόρους και όπως είπα προηγουμένως ο Στόλωτος αυτή τη στιγμή ελέγχει ποια είναι αυτά τα είδη τα οποία είναι σε αυτή την περιοχή και είναι στο συμφέρον μας αυτή τη στιγμή την ταχεία εισαγωγή ενισχύει αυτή τη σύμβάση, καθώς επίσης και ε, την πλήρη εφαρμογή όλων εκείνων των διατάξεων τα οποία θα είναι δεσμευτικά για όλες τις χώρες, για τους συμβαλλοντών, ώστε το, ο στόλος μας αυτή τη στιγμή σέβεται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι δεσμευτικά, είναι προσωρινά Αυτά είναι εθελούσια μέσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε εμείς να μετατρέψουμε όλα αυτά τα μέσα τα οποία υπάρχουν, αλλά δεν, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο με όλους τους συμμετέχων εκ μέρους όλων των συμμετοχών, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν οι νέες οι οργανώσεις προσπαθούν με πλήρη προσπάθεια και πλήρη ταχύτητα να εφαρμόσουν αυτά τα νέα μέτρα τα οποία έχουν καθομολογηθεί και κατά αυτόν τον τρόπο να φτάσουμε στο, επιθετικό, στο επιθυμητό εκείνο σημείο το οποίο θέλουμε. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή σα έδειξα ποια είναι η δική μα δέσμευση, ποια είναι η δυνατότητα μετατροπή αυτή. Όταν τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να υπάρξουν και τροποποίησεις οι οποίες θα πρέπει οι, οποία, οι τρεις έρχονται από τρεις παράκτιες χώρες και τρεις τροποποίησεις από μη παράκτητες χώρες. Όλα αυτά έχουν επικυρωθεί και για τα Φάρουερ, η Δανία, η Κούβα έχουν εγκρίνει. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε πως θα υπάρξει ένα άλλο παράδειγμα της δικής μας παρουσίας εκεί εάν θα θέλαμε πραγματικά να έχουμε την τάχη ε, επικύρωση αυτή της σύμβασης και αυτό θα είναι σε ε, πλήρη εφαρμογή σεβόμενη εκείνα τα είδη τα οποία θα πρέπει να προστατευτούν. Είμαι εγώ στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση που θέλετε να θέσετε. Ευχαριστώ. Ε, Τώρα θα λάβω εγώ το λόγο που είμαι η συγγετρία. Διάβασα έτσι στα πρόχειρα την ε, πρόταση για αυτή την σύμβαση και να σας πω πρώτα πρώτα κάτι γενικού χαρακτήρα για τον ειρηνικό. Ισχύει το ότι έχουμε τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα ίδια αυτά τα οποία δίνουν να δυνατότητα στα πλαίσια της εφαρμογής αυτών των συμβάσεων να εξαιρούνται κάποιες ζώνες που αφορά τα λιγότερο μεταναστευτικά είδη. Για ανοιχτή θάλασσα μιλάμε. Όμως, εξαρτάται τι, τι, τι μέτρα διατήρησης γίνονται και ισχύουν για διατήρηση και διαχείριση από τα παράκτια κράτη. Οπότε, γενικώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον ελληνικό, όπου μεγάλες περιοχές ανήκουν στην επικράτεια κάποιων κρατών, των παρακτήων χωρών, διαπιστώνω ότι για κάποια είδη τα οποία είναι πάρα πολύ μεταστευτικά, έχουμε αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν για την εκτή θάλασσα και όχι για τα χωρικά είδατα κάποιων χρόνων μελών. Γι' αυτό και σας λέω. Αυτό είναι γενική παρατήρηση. Επομένω, ισχύουν γενικέ αρχέ του δικαίου, γιατί εδώ πέρα μιλούμε για αυτά τα άκρο δραστηριστικά επίση. Κάτι το οποίο έλκυσε την προσοχή μου. Δεν ξέρω αν είναι δική μου προσωπική ερμηνεία το, του ότι παρά το το άρθρο 7 της σύμβασης του ΟΗΕ που αφορά αυτά τα είδη τα αλληλεπικαλυπτόμενα. Πρόκειται για κάποιου περιφερειακούς οργανισμούς ανοιχτή θάλασσας που έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν για αυτά. Δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 4 τα παράκτια κράτη είναι δυνατόν πολλές φορές να αναστέλουν την εφαρμογή κάποιων μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών για τα χωρικά του ύδατα. Αυτή είναι δική μου ερμηνεία. Αν θέλετε το συζητάμε. Βεβαίω. Ακριβώ επειδή έχει και η την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να προσχωρήσει μια τέτοια σύμβαση. Και ελπίζουμε ότι όπω και εμεί θα δείξουν το ίδιο πνεύμα συνεργασία και τα παράκτια κράτη. Όπω και έχουν τα πράγματα. Ε, για να δούμε. Πόσα σκάφη έχουμε στον ελληνικό. Δύο πολωνικά νομίζω. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε και στόλους από άλλα κράτη-μέλη. Μήπως μπορείτε να μας ε, διευκρινίσετε. Αυτά είχα να σας πω. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι φυσικά για την νέα ε, πόδα, Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της πόδα. Και βεβαίως περιγράφεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. αν κανείς αποφύγει τη διαδικασία της συνένεσης και υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό ε, βήμα για να έχουμε ένα σύγχρονο RFMO, ε, ΠΟΔΑ, Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης Αλίας. Η Χιλή αλλά και άλλες αμερικανικές χώρες έχουν επικυρώσει. Είπατε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση στα μέτρα διαχείρισης. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι όταν ε, αλλιεύονται κοράλια ή σφουγγάρια ε, υπάρχουν όρια ας πούμε 30 ε, κιλά για τα σφουγγάρια και 20 για τα κοράλια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 100 κιλά ανατόνο κλπ. Δεν ξέρω αν τούτο αλλάζει μετά την επικύρωση αυτής της ποδά. Και το τελευταίο σχόλιο, είναι περισσότερο σχόλιο μάλλον δεν είναι ερώτηση, αφορά στις ιστορικές αλλιεύσεις σε αυτή τη συγκεκριμένη RFMO, ε, την ποδά. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Στόλη αλλιεύουν στα ανοιχτά της χιλής για το ε, σαφρίδι Αυστραλίας, Jack Mackerel. Και ε, δυστυχώς όμως αυτή η κατηγορία ψαριών, μάλλον αυτή η αγορά, σχεδόν κατέρευσε. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε την ευθύνη του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το φαινόμενο. Ζητώ συγγνώμη που δεν θα μπορέσω να παραμείνω εδώ μέχρι το τέλος, θα μείνει όμως ε, συνεργάτης μου, διότι πρέπει να πάω και σε άλλη συνεδρίαση. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω στα γενικά σχόλια. Πρόκειται για μια σύμβαση για, ε, για την ανοιχτή θάλασσα Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επισημάναμε ότι μας ενδιέφερε επίσης η διαχείριση των βασικών αλληλεπικαλυπτόμενων ειδών. στην ανοιχτή θάλασσα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει το άρθρο 4 περί συμβατότητες και τα αναγκαία μέτρα περί συμβατότητες, ε, που και αυτά είναι σύμφωνα με τη Συμφωνία της Νέας Υόρκης και ίσως αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες αυτής της σύμβασης. Στο άρθρο 20 για την υιοθέτηση μέτρων συντήρησης προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής και υιοθέτησης και εφαρμογής μέτρων ε, για τα αλληλεπικαλυπτόμενα είδη αλλά και για τα EEZ. Γιατί οι παράκτιες χώρες επέμεναν να υπάρξει η Σύμβαση Ανοιχτή Θάλασσας αλλά έπρεπε να προβλεφθεί και το τι θα συμβεί με, τους, με τα αλληλεπικαλυπτόμενα είδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα στη σύμβαση και εμείς το εκτιμούμε αυτό ιδιαίτερος γιατί επιμείναμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κυρία Πρόεδρε, εσείς ρωτήσατε για την παρουσία μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία σκάφη. Δύο εξ αυτών είναι πολωνικά, το ένα είναι ολλανδέζικο. Η κυρία Λοβέν ρώτησε και απαντώ όλες οι παράκτιες χώρες της Λατινικής Αμερικής συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις από την Κολομβία στο Περού, την Χιλή, το Εκουαδόρ. Και ανέφερα τις χώρες που επικύρωσαν. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν είναι μεταξύ εκείνων που επικύρωσαν τη σύμβαση, ωστόσο. Τώρα, ως προς το τελευταίο σχόλιο που έκανε η κυρία Λοβέν, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε εντός της σύμβασης, αλλά υπάρχει και μια ένα ενδιάμεσο μέτρο που εγκρίθηκε τρεις φορές μέχρι τώρα για τους, τα αλληλεπικαλυπτόμενα είδη και πιο συγκεκριμένα το μαυροσάφριδο Αυσταραλίας, θα υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση ε, στο άμεσο μέλλον. Θα σταματήσω εδώ κυρία Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και περαιτέρω δυνατότητα συζήτησης αυτής της σύμβασης και δεσμεύεται και η Κομισιόν ότι θα προχωρήσει το ταχύτερο στην επικύρωση ε, αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Ναι, Πολύ σύντομο ερώτημα. Ξέρετε πότε η Χιλή θα υπογράψει και θα επικυρώσει τη συμφωνία αυτή. Μάλλον υπέγραψε, αλλά πότε θα επικυρώσει. Όχι, δεν έχω αυτή την πληροφορία. Έλεγαν ότι θα την επικυρώσουν πολύ γρήγορα και είναι προς το συμφέρον τους. Διότι είναι και η βασική χώρα ε, αλίας Είναι πως τους ενδιαφέρει να το επικυρώσουν το ταχύτερο δυνατό. Αλλά δεν έχω την πληροφορία ακόμα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Παρουσίαση της έκθεσης θα γίνει σύντομα. Δεν ξέρω σε ποια ακριβώς συνεδρίαση, ωστόσο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σεσάρη και έτσι κλείνουμε και με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και ερχόμαστε στο σημείο 12, το οποίο έχει πάει στο απόγευμα. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 13, που είναι η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Έχουμε την κυρία Ράιμεν, Ράιμερς, το ε, σχέδιο προϋπολογισμού συζητήθηκε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ράιμερς. Θα ακούσουμε από την Κομισιόν. Κυρία Ράιμερς, τι θέλετε, να μιλήσετε πρώτη ή να μιλήσει πρώτα η να μιλησει πρωτη Ωραία, ας ακούσουμε πρώτη την Κομισιόν. Thank you, Madam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Αυτό που προτείνω αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε μια παρουσίαση σύντομη στι 20 Απριλίου διπλωθεί από την Κομισιόν και να κάνουμε μια μικρή σύντομη παρουσίαση. Και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να τοποθετήσω πού βρίσκεται ο προπολογισμό. Είναι ο δεύτερο προπολογισμό υπό το καθεστώ τη Λισαβόνα και είναι πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά όσον αφορά τη διαδικασία του προπολογισμού. Είναι 20 χρόνια που δουλεύω στον το καθεστω τη Λισαβόνο και είναι η δεύτερη χρονιά πραγματικά όπου δεν υπάρχει οθετηθεί ακόμα προπολογισμό και η κατορθώσαμε τότε να τον ευθετήσουμε πριν από το τέλος του χρόνου, ενώ δεν είχε γίνει νωρίτερα, το είναι η δεύτερη, ο δεύτερος προϋπολογισμός υπό τη Λισαβόνα, ε, επαναλαμβάνω, και γνωρίζει η Επιτροπή σας ότι θα έρθει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή με προτάσεις όσον αφορά το πλαίσιο ε, για ένα πολιετές σχέδιο στις 29 Ιουνίου. Νομίζω αυτή τη στιγμή το καλύτερο που, που μπορούμε να κάνουμε, αυτό το οποίο ο κ. Πίτρο όταν υιοθετήθηκε ο προπολογισμό, όταν χαρακτήρισε τον προπολογισμό, ότι είναι μια λεπτή, λεπτεπίλεπτη ισορροπία όσον αφορά την ανάπτυξη και υπάρχουν 500 εκατομμύρια, ε, για, για 500 εκατομμύρια Ευρω, Ευρωπαίους. Έτσι όπω παρουσιάστηκε ο προπολογισμό ήταν σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη, και θα, πρέπει, θα έπρεπε να διατηρηθεί η ισορροπία για την ανάπτυξη αλλά και τις διαπάνες που θα έπρεπε να γίνουν υπό αυτά το καθεστώς και βεβαίως θα πρέπει να επικρατήσουν όλα αυτά σε όλες τις χώρες μέλη. Για να σας δώσω ένα, μια ιδέα από όλα αυτά γι' αυτά πρότεινε η Κομισέ 145 εκατομμύρια δις τα οποία δίνονται και υπάρχει μια αύξηση 27% σε αυτό το θέμα αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τροπολογία η οποία προτείνεται είναι 132 ε, δις όταν συγκριθούν βεβαίω όλα αυτά με τα προηγούμενα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο έχονται υπόψη αυτή, όλα αυτά τα θέματα, εφόσον υιοθετήθηκαν το τελευταίο χρονιά, θα πρέπει να υπάρχουν οι ε, δαπάνε οι οποίε έχουν προβλεφθεί και οι οποίε θα πρέπει να δώσουν, έδωσαν μια συμβαστική λύση για την αύξηση. Και η αύξηση κατά 2,9% για τον από τον προϋπολογισμό του 2010. Εάν δούμε πραγματικά τον τίτλο 11, το κεφάλαιο 11, το τι συνέβη αυτή τη στιγμή με τον προϋπολογισμό. Οι αριθμοί που υπάρχουν είναι ένα δις ευρώ για τις δαπάνες, προβλεπόμενες δαπάνες οι οποίες υπάρχουν από τα, από τα 98 δις τα οποία υπάρχουν. Και αν τα συγκρίνουμε μεταξύ του 10 και του 11. Βλέπετε ότι είναι πραγματικό, έχουμε το αυτό ύψος ποσών τα οποία υπάρχουν για τον προϋπολογισμό με μία ελαφρή αύξηση. Οι πληρωμές, οι δαπάνες πληρωμές οι οποίες θα γίνουν 78 798 δις ευρώ. Αυτό το οποίο προτείνω αυτή τη στιγμή είναι να περάσουμε τα διάφορα κεφάλαια του προπολογισμού και να υπενθυμίσω ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του προπολογισμού ε, πώς έχουν κατατμήματα. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω θα το πάρω κατά, κατά σειρά προ, όχι προτεραιότερα σημασία οι οποίε έχουν και βάρο και έχουμε ένα προπολογισμό αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια μάζα ποσών τα οποία και αφορά βεβαίω και την αλληλεία. Και, και εκπροσωπεί τα δύο-τρία από τις ε, δεσμεύσεις υποχρεώσεων που έχουμε αναπτύξει αυτή τη στιγμή. Αυτά τα οποία προτείνονται 672 εκατομμύρια είναι 2,2 αύξηση του προπολογισμού σε σχέση αυτό από το 10 στο 11. αυτό αυτός μέσο είναι ένα πάρα πολιτικά εργαλείο και αυτό είχε οριστεί στην αρχή της ε, αρχές της εποχής και βεβαίως υπήρχε μια προσπάθεια προγραμματισμού όλη αυτή μέσα στα χρόνια γι' αυτό και ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει για τα κράτη-μέλη και βεβαίως όταν η Κομισιό ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει υποβληθεί εκ μέρου των κρατών μελών προσπάθησε να δώσει μια συνολικό ποσό το οποίο είχε προβλεφθεί σε αυτό το κεφάλαιο σε όλη την πενταετή περίοδο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλος αυτοματισμός, αν θέλετε, όσον αφορά την καθέτος εφαρμογή. Όσον αφορά τις δαπάνες πληρωμών, σε αυτό, το, σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται όχι μόνο αυτά, αλλά και έκτακτες ε, δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τις οδηγίες ε, ε αλλιευσής που ξεκίνησαν από το 2006. Είναι 540 δις και υπάρχει μια αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Το 12 λοιπόν πιστεύουμε ότι στο EFF θα πάρει μεγάλη ταχύτητα, κανονική ταχύτητα και θα φτάσουμε στο ποσό το οποίο έχουμε προβλέψει και αυτή την, την περίοδο και θα δούμε 30 εκατομμύρια τελικών πληρωμών από το κλείσιμο των ε, πληρωμό που θα πρέπει να γίνει μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Δεύτερος τομέας πολύ σημαντικός πληρωμός αυτής της πολιτικής είναι η διεθνή αλίευση σε ανοιχτέ θάλασσες. Αυτό εκπροσωπεί το 60% των δικών μας δαπανών και επινάμε βεβαίω για τα ποσά εκεί τα οποία έχουν προβλεφθεί για τις συμφωνίες ε, εταιρικέ συμφωνίε που έχουν προβληθεί με διάφορε χώρε. Επίση, μιλάμε για τα ποσά οικεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε αναχείρα για να εκπληρώσουμε τι συμφωνίε εκείνε που έχουμε για τι περιφερειακέ αλλιευτικέ συμφωνίε. Και βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει ρευστό σε αυτό το θέμα. Σε προσθήκη σε όλα αυτά, επίση, κάνουμε μια θελούσια συμβολή η οποία θα μπορούσε να έχει εκείνη σε αυτό το τομέα. Και βεβαίω ο προπολογισμό δεν μπορεί να καλύψει όλου αυτού του τομέε δραστηριότητα οι οποίοι προβλέπουν και υπάρχουν ακόμη μικρά ποσά τα οποία έχουν προβλεφθεί για, για για το δικαστήριο της, ε, για το δίκαιο της θάλασσας. Νομίζω πως πραγματικά είναι πολύ σταθερό αυτό το πράγμα όσον αφορά το 11 και όσον αφορά τις δαπάνες πληρωμών προβλέπουμε 154 εκατομμύρια, τα οποία είναι σχετικά μικρή αύξηση με την προηγούμενη χρονιά. Βεβαίω, η ιδιαιτερότητα αυτού του προπολογισμού είναι ότι υπάρχουν μερικέ δαπάνε οι οποίε βρίσκονται στο κεφάλαιο αυτό και τα άλλα είναι στο αποθεματικό. Και βεβαίω αυτό είναι ο βασικό άξονα ο οποίο υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο ε, κεφαλαίων. Το επόμενο, κεφάλαιο σε σημασία είναι αυτό που άπτεται όσον αφορά τον έλεγχο. Τον έλεγχο του και είναι το κεφάλαιο 8 και βεβαίω υπάρχουν τρεις διαφορετικές δαπάνες οι οποίες καλύπτονται. Τα προγράμματα των κρατών για τον έλεγχο, μέτρα τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν οι χώρε όσον αφορά την εφαρμογή τη κοινή αλληλευτική πολιτική και βεβαίω θα υπάρξουν εκεί δαπάνε, καθώ επίση και με την εισαγωγή σε εφαρμογή των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων χωρών, τι ευθύνε που οποίε θα λαμβάνει η χώρα σε αφορά τι ανταλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη νέα τεχνολογία για την παρακολούθηση των, των στοιχείων ε, πληροφορική σε εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την αποβίβαση και εκφόρτωση. Έτσι λοιπόν συμβα... Ε, ε, εμείς πάρα πολύ για τους 12 όσον αφορά τα κράτη-μέλη και την αύξηση της δικής του ηλεκτρικού του ηλεκτρικού μηχανισμού και και θα διαδεθούν 47,5 εκατομμύρια για αυτό το σκόπο, στο σκοπό. Επίσης, προποτείνουμε να μείνουμε στα 2,3 εκατομμύρια για αυτό το θέμα. Επίσης στο Βίγκο υπάρχει μια ελεκτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα και βεβαίω θα πρέπει αυτή να είναι σε ευθεία γραμμή με το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα. Το επόμενο κεφάλαιο είναι όσον αφορά το οποίο καλύπτει τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από τα προγράμματα που έχουν τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Και βεβαίως θα πρέπει εδώ να υπάρχει μια επιστημονική πληροφόρηση που θα πρέπει να δοθεί. Και βεβαίως εδώ με μια αύξηση που θα πρέπει να υπάρχει 4,1% όσον αφορά τις δαπάνες πληρωμών και θα φτάσουμε σε 42 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως όσον αφορά την αγορά αλλίας, σε αυτό το τομέα καλύπτεται την κοινή αγορά, ε, την, αγορά, την κοινή αγορά η οποία υπέρχεται αυτά τα λέματα και καλύπτει επίση τα προγράμματα εκείνα τα οποία υποστηρίζουν ε, αυτούς οι οποίοι έμπρακτα δουλεύουν εκεί και τους διάφορους πράκτορες για αυτό το τομέα. Προβλέπετε λοιπόν ποιο είναι το ποσό το οποίο υπάρχει αυτούς κάθε χρόνο και υπάρχει μια σταθερότητα και μιλάμε για 30 εκατομμύρια για δεσμεύσεις και για πληρωμές έχουμε μια αύξηση για μέχρι 30 και έχουμε 27 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το θέμα. Υπάρχει, υπάρχει ένας ακόμη ε, κεφάλαιο, το 4, το οποίο είναι της διακυβέρνησης της Αλίας και βεβαίως με, υπό αυτό το κεφάλαιο δίνουμε εκείνε τι παραχωρήσει και επιδοτήσει που δίνουμε στι διάφορε περιοχέ για την Αλία, σε αυτέ οι οποίε συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία που έχει γίνει με, μεταξύ των περιφοριών. Και βεβαίω είναι οι διαλέξει, τα περιοδικά, οι δημοσιεύματα τα οποία γίνονται για αυτό το θέμα και νομίζω αυτό μεταξύ υπάρχει 6 εκατομμύρια, 4,4 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Περαιτέρω θα ήθελα να σα μιλήσω για μια ακόμη πολιτική. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Έχουμε προτείνει την διαδικασία συναπόφαση για αυτά τα θέματα και σύμφωνα με, τη, με τις αρχές αυτές προτείναμε το 12 μπήκε αυτό το ποσό το οποίο είχε προβλεφθεί μέσα 6,6 εκατομμύρια όσον αφορά τις δεσμεύσεις. Βεβαίως αυτές οι προτινόμενες δεν μπαίνουν στον προπολογισμό όπως γίνεται όπως για τις συμφωνίες των άλλων των αλληλευτικών συμφωνιών που έχει γίνει. Μπαίνουν απλώς στο αποθεματικό. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο το παρουσιάζουμε εδώ. Είδου λοιπόν ποια ήταν η συνολική σφαιρική παρουσίαση Βλέπετε λοιπόν τι προτείνεται όσον αφορά τα θέματα της αλληλείας, μια σφαιρική και ε, αντιμετώπιση των θεμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε ε, Τζόναθαν. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ εμπεριστατωμένη η παρουσίαση. Μερικές φορές είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όλους αυτούς τους αριθμούς, καθώς δεν ασχολούμαστε σε καθημερινή βάση με αυτούς. Πράγματι, περνά, ζούμε σε δύσκολες εποχές. Οι χώρες μέλη πρέπει να καταβάλουν τεράστια ε, προσπάθεια και να βρουν και μία μέση λύση για να διατηρηθεί η αλληλεία ως πηγή εσόδων στην Ευρώπη. Ενώ από την άλλη πλευρά πρέπει να διατηρηθούν τα ηχθή αποθέματα και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντανακλάται στο πλαίσιο του πολιετούς ε, χρηματοοικονομικού πλαισίου. Ε, πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του κλάδου και των εμπλεκομένων. Και στη συνέχεια να υπάρξει ένα follow-up και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Όσον αφορά το EFF, αυτό λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία και αυτού το αντανακλάται και στον προϋπολογισμό. Απαιτούνται έλεγχοι να είμαστε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι ο έλεγχος και η επιτήρηση αποτελεί τμήμα της κοινή πολιτικής αλίας. Ούτως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην υπάρχουν παρεκτροπές. Αυτά είναι τα αρχικά μου σχόλια και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την συνεισφορά. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέντεκ θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποφεληθώ <coughs> της παρουσίας της Κομισιόν για να κάνω μια ειλικρινή πρόταση. Θα ήθελα να προτείνω ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να ε, παρακολουθήσουμε τις την τεχνολογική εξέλιξη ώστε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη αλληλεία ε, με, κάνοντας παράλληλα τις απαραίτητες ε, οικονομίες. Ως προς την ηλικία των σκαφών γνωρίζουμε ότι είναι πεπαλαιωμένα. Ο μέσος όρος, είναι πάνω από 20, μέσος όρος ηλικίας πάνω από 20 έτη. Ως προς τις σε σχέση μάλλον με τις κλιματικές αλλαγές, επίσης θα πρέπει να έχουμε μια βιώσιμη αλληλεία ε, που θα λαμβάνει υπόψη την ε, ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητα για μας. Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει και στην μείωση των ε, αερίων διοξιδιού του άνθρακα. Ε, έχει να κάνει με κατασκευή σκαφών που όχι, δεν θα λιεύουν περισσότερο, αλλά θα λιεύουν καλύτερα ε, δαπανώντας λιγότερα. Αν λοιπόν ε, συμφωνείτε, θα ήθελα να καταθέσω αυτό το πιλωτικό σχέδιο εξ ονόματος της Επιτροπής Αλίας, ε, ούτως ώστε να υπάρξουν και άλλες προτάσεις και να προχωρήσει αυτό το πιλωτικό σχέδιο. Αυτό ήθελα να σας προτείνω. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Ρόντουστο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπλήσωμαι, για να είμαι ειρικρινής, Αλλά στο αφήσω αυτό, κατά μέρος. Έχω τρία ερωτήματα προς τον κύριο Τζάνσεν. Καταρχήν, το 2011 είχαμε μια αύξηση στο κεφάλαιο 3 για τον φορέα ελέγχου. Τότε λέγαμε ότι ο φορέας ελέγχου θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει και στα διεθνή ύδατα. Δεν είναι απόλυτα σαφές για ποιο λόγο ε, η Κομισιόν μείωσε αυτό το ποσό, διότι ήταν πολύ σημαντικό για να ελέγχεται η πλεονασματική αλληλεία σε αυτές τις περιοχές. Εμείς εδώ στην Επιτροπή Αλίας ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ως προς τους ε, πόρους EFF. Για ποιο λόγο υπάρχει μείωση εκεί. Και επίσης, τι γίνεται με το θέμα της συγχρηματοδότησης των ελέγχων που γίνονται σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Νομίζω ότι ε, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτό το μέτωπο και να μας δω, εξηγήσετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μείωση. Η Πρόεδρος. Έχω κι εγώ κάποια σχόλια προς τον κύριο Τζόνστον. Είπατε ότι η αύξηση των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων έφτασε στο 3,7. Εγώ βλέπω στο κεφάλαιο 3,1. αλλά αν αφαιρέσουμε τα 16,6 εκατομμύρια για ναυτιλιακή πολιτική, που δεν είναι αλληλευτική πολιτική, η ουσιαστική αύξηση είναι 1,4% και αυτό για μένα είναι συγκητικό. Διότι η αύξηση της ε, αύξηση των κονδυλίων για την πολιτική αλίας είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις αυξήσεις σε άλλες πολιτικές. Και ουσιαστικά μέσα σε ένα-δύο χρόνια θα ξεπεραστεί εντελώς. Δεν ξέρω, ότι, δεν ξέρω αν υπάρχει οποιαδήποτε δικαιολογία επ' αυτού. Δεύτερον, υπάρχουν δύο σημαντικές γραμμές του προϋπολογισμού που θα πρέπει να αυξηθούν το 1107 για την διατήρηση, είναι το 1 και υπάρχει ο συγκεκριμένος στόχος υπαριθμών 3 για την διασφάλιση της βιωσιμότητας και της εφικτότητας των γερμανικών αποθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική άποψη Νομίζω ότι το κεφάλαιο αυτό απαιτεί περισσότερη χρηματοδότηση, διότι εδώ υπάρχει η πιθανότητα να περιληφθούν κάποια projects τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στο EFF. Και έτσι θα βελτιωθεί η επιστημονική βάση για να έχουμε καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων στην Ευρώπη. Κάτι πάρα πολύ, ένα θέμα πολύ σύνθετο η Κομισιόν επιμένει ότι το 2015 σε όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα αποθέματα θα πρέπει να έχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Πώς θα επιτευχθεί αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Ρέιμενς ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση του 1107, της γραμμής 1107 και υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε έναν από τους στόχους που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μια άλλη γραμμή που επίσης είναι σημαντική είναι η 1108 για τον έλεγχο. Ιδιαίτερα επειδή η Κομισιόν ε, προβλέπει για το προσεχές έτος κάποια προγράμματα που είναι πρώτης προτεραιότητας, προγράμματα ας πούμε λασιμότητας και άλλα. Ε, Εκπλήσωμε λοιπόν που δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση διότι ε, ο φορέας ελέγχου ουσιαστικά, μάλλον η χρηματοδότηση για τον φορέα ελέγχου μειώνεται από 9,1 σε 2,7 εκατομμύρια. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν γιατί εισάγεται αυτή την μείωση. Ε, ε, για ποιο λόγο πλήττεται τόσο σκληρά αυτός ο φορέας αυτή η υπηρεσία ελέγχου. Ε, ε, να πω και κάτι έτσι διαφορετικό. Εξεπλάγην ε, για την εξεπλάγει από τους υπολογισμούς που έγιναν σχετικά με την αλία. Ωστόσο, στις εξηγήσεις που δώσατε είπατε ότι προβλέπετε ότι ενδεχομένως να υπάρξει συμφωνία με τη Σενεγάλη. Αλλά αυτό είναι κάπως περίεργο διότι ε, ποτέ δεν ξέραμε ότι θα επιστρέψουμε σε μια συμφωνία με τη Σενεγάλη, μια συμφωνία που έχει εκπνεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό είναι πολύ περίεργο. Το λέω αυτό έτσι, σε παρένθεση. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Ρέιμεν σχετικά με την μείωση από 3,1 σε 1,4. Κοιτάξτε, η πολιτική ναυτιλίας δεν είναι ε, οπωσδήποτε αλλιευτική πολιτική. Ίσως υπάρχουν κάποιοι λόγοι, αλλά θα ήθελα να μάθω ακριβώς ε, περί τίνος πρόκειται. Και σίγουρα θα κατατεθούν τροπολογίες σχετικά με τις γραμμές 11.07 και 11.08. 8. Κύριε Τζόνσον, έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση από την κυρία σε σχέση συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων η οποία θα πρέπει να γίνει είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά και να υπάρξει πραγματικά μην υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο μπορεί να πτυχθεί και το οποίο να το μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε σε αυτή τη φάση. Πιστεύω πως η Κομισιόν είναι ανοιχτή σε προτάσεις που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίω σε σχέση με το πρόγραμμα για την προετοιμασία υπάρχει μια διαδικασία η οποία έχει εισαχθεί και αυτή βεβαίω θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Θα ανακοινωθεί η διαδικασία και βεβαίω όταν η Επιτροπή θα δώσει τη δική τη άποψη προ το Γενικό Εισηγητή για αυτό το θέμα και τι προπαρασκευαστικέ εκείνε διαδικασίε οι ε, οποίε χρειάζονται ω αναφορά για αυτό το Συμβούλιο για τα πιλωτικά προγράμματα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να απαντηθούν τα τα πιλωτικά εκείνα που προτάθηκαν από τον κύριο Πάλα. Και το μόνο που θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω για αυτά τα πιλωτικά είναι ότι η ιδέα χρησιμοποιήσεως για την ευρωπαϊκών κεφαλαίων για, ε, ε, για το κτίσιμο πλοίων δεν νομίζω πως πρέπει να έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο και δεν νομίζω πραγματικά ότι αυτό θα υπάρξει μέσα στις προοπτικές της Κομισιόν στο μέλλον. Όσον αφορά τις ειδικέ ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν, όντως η τα πρακτορία ελέγχου, οι εταιρείε ελέγχου έχουν μια αύξηση όσον αφορά ε, το ποσό αυτό στον προπολογισμό του 11 και του 12 και βεβαίως αυτό το ελέγχει η Κομισιόν και αυτό το Κοινοβούλιο ψήφισε μία αύξηση όσον αφορά αυτούς τους ελεκτικούς μηχανισμούς και είναι πάνω από αυτό το πρόγραμμα και όταν εμείς θα επανέβουμε πέρσι για αυτό το θέμα διασαφηνίσαμε και πιστεύουμε πως τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα για τις εταιρείε εκείνες, για αυτή την εταιρεία η οποία έχει υπογράψει διάφορες συμφωνίες όσον αφορά τα, τα σκάφη και τα πλοία και θα πρέπει να δούμε με βάση αυτή την αρχή οι χώρες εκείνες οι οποίες θα θέλουν να έχουν ηλεκτρικούς μηχανισμό τι σημαίνει έλεγχος αυτό και πώς μπορούν να συνεργαστούν, ποιος παίγει αυτές τις διαστηριότητες ελέγχου και το πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή για την υπάρξει αυτή η αύξηση στον προπολογισμό είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε πως για να, κατα... για να δαπανηθεί τέτοιο μεγάλο ποσό ότι είχαμε αρκετές εκτιμήσεις που... και αρκετές αναλύσεις οι οποίες υπάρχουν στον αφορά όλη αυτή την κλιμάκωση και όλη αυτή την διακλάδωση που υπάρχει στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να έρθουμε πίσω ξανά στο σχέδιο χρηματοδότηση, αυτό το οποίο προβλέπεται όσον αφορά την εταιρεία ελέγχου αυτή που υπάρχει σε αυτό το θέμα και όπως συνέβη πέρσι θα συμβεί και φέτος και αυτό βεβαίως είναι το προνόμιο της ε, από το του προπολογισμού που μπορεί να εισάγει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη τώρα, καθώς επίσης και την άσκηση του ελέγχου εκ μέρους αυτό και τη συγχρηματοδότηση, ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρξει, αν αυξηθεί το ποσό το οποίο υπάρχουν κατά 2 εκατομμύρια ευρώ και για τον φάκελο το οποίο υπάρχει είναι περίπου της τάξης στο 4%. Είναι πολύ πιο ψηλά από το μέσο όρο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στα κράτη-μέλη και βεβαίως εφόσον έχουμε αυξήσει φέτος αυτό το ποσό τη συγχρηματοδότηση που γίνεται και εκπροσωπεί βέβαια το 90% του κόστους αυτή η συγχρηματοδότηση που προβλέπεται και η οποία έρχεται εκ μέρους της Κομισιό. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κρατη μελη θα συνεχίζουν να ασκούν αυτό το έλεγχο ο οποίο επιβάλλεται. Το ερώτημα το, το οποίο από την κυρία Φράγκα σε σχέση με την αύξηση για την Ελλιάνα δεν είναι 3,1% είναι κάτι λιγότερο. Βεβαίως μιλάμε εδώ για τον προπολογισμό στι στις υπόθεσεις του θαλασσίου, του προϋπολογισμού ε, είναι, είναι πολύ λιγότερο από το 3,1 εάν εξάγουμε αυτά τα οποία έχουν σχέση με το θαλάσσιο τομέα και είναι πολύ λιγότερο. Βεβαίω, ε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το ένα τομέα πιο κοντά στον άλλο και τον τρόπο αυτό μπορούμε να δούμε ο, να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός όσον αφορά τις υποθάσεις, καλύτερη γνώση, καλύτερη ανάλυση που άπτεται της αλίας και όλα αυτά μπορούν να διευκολύνουν την οικονομική βιωσιμότητα της αλίας γενικότερα. Τούτων λεχθέντων 1,3% είναι πολύ λιγότερο αλλά εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή δύο πράγματα ακόμη. Ένα είναι ότι όπως το EFF και τα άλλα διαφορετικά ταμεία έχουν ένα φυσικό πρόγραμμα όσον αφορά το θέμα αυτό και αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή του προπολογισμού. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε εμείς να έχουμε μια αύξηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η γενικότερη αύξηση είναι 3,4% αλλά υπάρχουν ειδικοί τομείς του προπολογισμού τα οποία έχουν υποστεί περικοπές και δεν νομίζω πως αρκούν αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό είναι μια δύσκολη επιλογή που θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν με τις παρούσες συνθήκες. Σε σχέση με, με το θέμα της έρευνας, βεβαίως εμείς έχουμε δεσμευτεί να πάρουμε αποφάσεις τον καλύτερο τρόπο, τρόπο με με επιστημονική τρόπο και έχουμε την καλύτερη διαδικασία αποφάσεως. Θα πρέπει να δούμε εκ του σύνοικες πάρα πολύ προσεκτικά ότι, και να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε λαμβάνεται είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το καλύψουμε. Και εάν υπάρχει ένα κενό συγνώση, τότε θα πρέπει να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να το καλύψουμε αυτό το κενό γνώση το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ευχαριστώ, κυρία. Πιστεύω πως δεν κατάλαβα καλά αυτό το οποίο έχετε να πείτε. Αυτό το οποίο ε, προβλέπετε για το 11 είναι ένας επιπλέον έλεγχος ο οποίος γίνεται σε διεθνή ύδατα. Ίσως δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι με τα κρατημέλη. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας έλεγχος πάρα πολύ σημαντικός, το οποίο μπορείτε να με διαφοροποιήσετε για αυτού του θέματος. Πρόεδρε, οι εξηγήσει οι οποίες εδώ μέχρι τούδε όσον αφορά την... Αυτό είναι κάπως πλασματικό η ένταξη δηλαδή στον προπολογισμό είναι όμως δική μας αρμοδιότητα. Είναι κάτι που σημαίνει, μάλλον κατά διάρκεια από την Ερμεριά Έχουμε το, το, τι, γίνεται, τι έγινε πέρσι και τι αλλαγές έχουμε επιφέρει όσον αφορά αυτές τις αλλαγές για τον προπολογισμό. Μια προς τον προπολογισμό ε, βασιζόμαστε πάντα στην προηγούμενη χρήση και στη συνέχεια έχουμε τις μεταβολές στον προπολογισμό. Ε, αλλά όμω όλα αυτά, όπω έλεγα πριν, γίνονται κάτι δεν είναι, είναι εικονικά κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι πραγματικά. Άρα για να δούμε τι γίνεται με την χρήση 11, τι αλλαγέ έχουν γίνει και τι ποσά αφορούν. Πρόεδρο, εγώ ε, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω. Πολιτική για τη θάλασσα, πολιτική για την αλία, γιατί αυτό το οποίο μα αφορά και πρέπει να δούμε εδώ πώ σχετίζουμε τα πράγματα και έχουμε και την επιστηστική βοήθεια. Οπότε δεν είναι θέμα λοιπόν για μας ε, τι γίνεται με την ε, ε, πολιτική που αφορά τη θάλασσα γενικά. Εμάς εδώ μας αφορά ακριβώς τι έγινε με την, με την ΚΑΠ. Έχουμε αυτό το 96% και έχουμε το 4% ε, οπότε αυτές οι περικοπές νομίζω ότι είναι θλιβερές και ο προπολογισμό είναι θλιβερός για αυτόν τον, ε, αυτό τον λόγο. Είναι δυνατόν να έχουμε με μια, ΚΑΠ και να έχουμε την άλλη μεριά ε, διαρθρωτικό ταμείο του ενός δις. δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στο ψυγείο η, η Αλία. Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε κάποια αύξηση όπως προτείνεται στον προπολογισμό. Γι' αυτό το 3,1% να υπάρξει προτεραιότητα γιατί εδώ έχουμε θέματα, έχουμε ελλείμματα. Τα ελλείμματα αφορούν την έρευνα και άρα θα πρέπει να μην γίνεται ουραγός η ελεία. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε επιστημονική ε, τεκμηρίωση γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Και όπως σωστά είπατε, αυτό είναι προνομίο του Κοινοβουλίου. Είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και εγώ ως μέλος της Επιτροπής Αλίας θα κάνω ό,τι μπορώ. Γι' αυτό λέγεται η την κυρία Ράιμερς. Οι προτεραιότητες θα πρέπει να τηρηθούν. Λάβετε υπόψη τι λέει ο προπολογισμό τη Γενική Διεύθυνσή σα. Γι' αυτό η κυρία Ρέιμερς θα πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή των ε, καταλήλων τροπολογιών. Έχετε το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως και καταλαβαίνω τον προβληματισμό της Επιτροπής σας θα ήταν περίεργο να μην καταλάβω, είναι δική σας αρμοδιότητα. Βεβαίως και μιλούμε για κατάρτιση του προπολογισμού. Εγώ σας παρουσιάζω την πρόταση του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπώ. Θεωρούμε ότι είναι εύστοχες οι προτάσεις μας όσον αφορά άλλε δαπάνε, λέμε εδώ πέρα ότι για εξωτερικέ δαπάνε όσον αφορά την αναπτυξιακή ε, βοήθεια έγινε περικοπή 70 εκατομμυρίων. 14,5 περικόπησαν από την ενίσχυση στι βιομηχανωμένε χώρε. Ε, από τον Γαλιλαίο, από τον κοπήκανε. Ε, εδώ πέρα νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μικρές περικοπές, Πενταροδεκάρε και γίνανε για βάσιμου λόγου Οπότε ξαναγυρίζουμε τώρα στο θέμα τη περιφερειακή υπηρεσία του Βίγκο. Όχι, η εντολή δεν επηρεάζεται από την πρικοδότηση. Η εντολή μένει ίδια. Και αυτό το οποίο έκανε, προσπάθησε να κάνει η υπηρεσία ήταν το να αναβλώσει ένα σκάφος το οποίο μέχρι τώρα με άμεσες πληρωμές ε, χρηματοδοτούσαν, επλήρωναν τα κράτη-μέλη. Αν θέλει τώρα αυτή η υπηρεσία να το αναβλώσει και του χρόνου και αν ο προπολογισμό παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, τότε τα κράτη-μέλη τα οποία ωφελούνται όσον αφορά το ότι εκπληρώνονται έτσι οι υποχρεώσει τους με τα FMO, τότε θα πρέπει να πληρώσουν για αυτά τα ποδά. Τώρα καταρχήν ο προπολογισμό με περισσότερη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Άρα θα αποκτήσει την κατάλληλη πρικοδότηση η υπηρεσία του Βίγκο. Όσον αφορά τώρα την πολιτική για τη θάλασσα, νομίζω ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ και τα συζητούμε, είπαμε ότι ουδέποτε έχει χρηματοδοτηθεί εκείνη η πολιτική εις βάρος της ΚΑΠ. Μιλάμε για αυτό το πολιτές πλαίσιο. Ε, η αλία το πιο σημαντικό ε, κεφάλαιο. Εκεί που καλύπτονται δαπάνες, γεωργίας, αλίας, υγείας, περιβάλλοντος και όπως κάθε τίτλος στον προπολογισμό έχει αυτό το οποίο ονομάζουμε περιθώριο που είναι ένα ποσό το οποίο έχει δεσμευτεί και το οποίο βρίσκεται και έχει ως όριο τέλο πάντων την οροφή που προβλέπεται για το οικείο κεφάλαιο. Νομίζω ότι απάντησα όσο μπορούσα καλύτερα για να σας καλύψω. Αν θέλετε διμερώς να τα πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πρότασή μας ως Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ρέιμερς. Η κυρία Ρέιμερς. Ασφαλώς πρέπει να συζητήσουμε όλες μας τις προτάσεις από κοινού. Και όλες οι εξηγήσεις Όντω υπάρχει εξωτερική πίεση, άρα θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην ζητάμε υπερβολικά πολλά και επομένως τελικά να μην φτάσουμε στο σημείο του να ζητήσουν άλλες επιτροπές περικοπές κατόπιν αυτής μας της, τακτικής. Άρα, επομένως, έτσι όπου είναι δύσκολη σημερινή συγκυρία, θα πρέπει να βρούμε έναν αλλακτικό τρόπο, να κάτσουμε και να αναλογιστούμε ποιες είναι οι κορυφές μας προτεραιότητες, ποιες είναι οι λιγότερο σημαντικές, αλλά βέβαια μια που είμαστε επιτροπή για την Ελία, θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τον, τον, την πρικοδότηση με αυτές τις προτάσεις και μετά να δούμε τι στρατηγική θα έχουμε στις διαπραγματεύσεις γιατί θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι επαφέ οι συζητήσει που θα γίνουν. Με μεγάλη μου χαρά ε, να, να, να μελετήσω τις προτάσεις σα, παρακαλώ τι εγγράφους και να προχωρήσουμε και να πρετανεύσει η λογική. Πρόεδρος, οπότε τώρα έχουμε την παρουσίασή σας που θα γίνει τον Ιούλιο, συζήτηση στην Επιτροπή και επίσης ε, το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις ε, τροπολογίες για τον προπολογισμό και όσον αφορά το σχέδιο της νομοδότησης που θα γίνει 18 Ιουλίου και η ψήφιση θα γίνει 31 Αυγούστου στην Επιτροπή μας. Σας ε, ευχαριστούμε. Κυρία Τζόνστον, πάμε τώρα στο 14ο σημείο. Ε, το 14ο σημείο αναβάλλεται γιατί το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε στο 15, σημείο 15, δηλαδή αποστολή την προσωπή τη Επιτροπή 13 με 16 Απριλίου, που πήγαν 10 βουλευτές εκεί πέρα. και η κυρία Πατραονέβες ήταν η επικεφαλής της αποστολής αυτής Νομίζω έχετε λάβει το σημείο της γραμματείας μας το οποίο σας ενημερώνει για το τι έγινε κατά αυτή την αποστολή. Τέλο πάντων. Ευχαριστώ τους πάντες. Ευχαριστώ την κυρία Πατράου. Το πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε κυρία Πατράου σας δίνουμε την σκητάλη ούτω ώστε να μας πείτε τα πιο βασικά από την αποστολή εκείνη. Έχετε το λόγο. Secretariado, eh, fico convicta και mesmo quem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 destas missões, eh, realmente Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι ε, κατά αυτή την, επίσκεψη μπορέσαμε να έχουμε επαφές πάρα πολύ κοντινές, αποτελεσματικές και να δούμε ε, πολλές πλευρές της ε, εκεί πραγματικότητας. Επομένως, για να έχουμε πολλές απόψεις ε, της πραγματικότητας έλεγα, είδαμε πολλούς, είδαμε και συνδικαλιστές, είδαμε και αλληλείς, είδαμε εκπροσώπους της ε, τοπικής ομοσπονδίας αλληλείων, ε, εκπροσώπους των πλειοκτητών, εμπόρους, βιομήχανους, συναντήσαμε πάρα πολλούς, ένα ευρύτατο φάσμα εκπροσώπων του κλάδου. Όμως συναντήσαμε και επιστήμονες ερευνητές γιατί προσπαθούμε να δούμε το θέμα του πόσο η βιώσιμη αλληλεία προϋποθέτει έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση. Επαφές επομένως σε υψηλό επίπεδο. Τον αρμόδιο υπουργό, γενικό διευθυντή εκπρόσωπους της τοπικής ε, περιφερειακής κυβέρνησης, τοπικές αρχές, ε, ακόμη και την ε, νομοθετική συνέλευση των Αζωρών. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η αποστολή. επισκέψεις, διαφορετικές χρονικές στιγμές. ανταλλαγή απόψεων. Και νομίζω ότι υπήρξε ειλικρίνεια, ήταν ε, ενδιαφέρουσες αρπαστικέ οι συζητήσεις μας. Και από τι δύο πλευρές. Νομίζω ότι ενδιαφέρθηκε έντονα ο, ο κλάδος και οι πρόσωποι του να μας ε, συναντήσουν. Υπήρξε επομένως, μπορούμε, πνεύμα ενθουσιασμού. εισηγήσει, παρουσιάσεις και επίση υπήρξε ευρεία συμμετοχή. Και επίση, και από δική μας πλευράς όλοι δουλέψαμε με ενθουσιασμό και όρεξη. Υπήρξε η παρουσία μας επομένως σοβαρή. Ήμασταν εκεί αυθεντικά παρόντες πραγματικά συμμετέσχαμε. Ε, είχαμε ένα σωρό ερωτήσεις που υποβλήθηκαν ε, παντού, σε κάθε επαφή. Και σας υπενθυμίζω ότι όταν πήγαμε να δούμε την τοπική συνέλευση, ήρθαμε σε επαφή με τους τοπικούς βουλευτές, την τοπική επιτροπή Ελίας, Και αυτό το οποίο αναδείχθηκε από τις επαφές μας ήταν ότι θα πρέπει διεξοδικά να συζητήσει το θέμα με ερωτήσεις για να προκύψει η εικόνα της πραγματικότητας. Είχαμε υποστήριξη επιμελητίας από την συνέλευση αυτή των Αζωρών και όσον αφορά την βιοπικιλότητα και όσον αφορά την πολλαπλότητα των επαφών είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις για την κοινή αλληλευτική πολιτική περιφερειοποίηση συμμετοχή των τοπικών περιφερειακών αρχών στην διαχείριση της αλίας. Επισημάθηκε το ότι η κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να μην χάσει από την ευελιξία της. Θα πρέπει δηλαδή η κοινοτική νομοθεσία να είναι με νομιόμορφη, αλλά να λαμβάνει υπόψη τις ιδιορυθμίες, τις ιδιομορφίες κάθε τόπο. Φυσικά και μιλήσαμε για το γάβρο τη Σαρδέλα, γιατί εδώ υπήρξε θέμα πιστοποίησης που προϋποθέτει αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικά μέσα για να καταπολεμηθεί η λαθρέα αλία, παράνομη αλία. Θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικέ οι τιμέ, να βρεθούν περισσότεροι αγοραστέ, θα πρέπει να αυξηθεί η πρώτη τιμή πώληση, να γίνεται καλύτερη απορρόφηση των πόρων από την κοινωνικά ταμεία, να βελτιωθούν οι υποδομέ. Γενικά πάντως θεωρήθηκε επιτυχής η συμβολή των κοινωνικών ταμείων από τις ε, κοινότητες των αλλιών. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα και σχέδια για την διεύρυνση δραστηριότητα με αλίευση ειδών που μέχρι τώρα δεν είχαν ιδιαίτερη αξία και επομένως ε, υπάρχουν άφθονοι σχετικοί αλληλευτικοί πόροι. να επίση επίσης διάφορα είδη διατροφής που έρχονται από την Αλία. που όπως τις Αζόρες είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούν οι αληφτικές κοινότητες της απότερης περιφέρειας. Έχουμε και κάποια εγκάρσια οριζόντια θέματα για όλα τα κρατημέλη, τα οποία επίσης ενδιαφέρουν όπως ας πούμε η υποστήριξη, η επιδότηση για τον εξυγχρονισμό του στόλου. Να μην ε, πολυλογώ, αλλά δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω όλους βουλευτές, ε, συνεργάτες, ε, διερμηνείς, την γραμματεία μας, γιατί κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες και για τη διοργάνωση της επίσκεψης αλλά θα πρέπει να τους ευχαριστήσω και για τα όσα έκαναν συμμετέχοντας εκεί. Διευκόλυνα το έργο μας. Και επαγγελματίες ήταν και πάρα πολύ συμπαθητική στάση τους. Άρα ήταν πολύ ευχαριστώ το κλίμα και έτσι όλα τα πρόβλεπτα ενός ταξιδιού μιας αποστολής μπορέσαμε να τα παρακάμψουμε. συμπαθάτε με για ό,τι τυχόν έγινε. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Νομίζω ότι έχετε όλοι λάβει αυτό το δισκάκι που περιέχει τις φωτογραφίες μας από τις εκδηλώσεις που έγιναν. Ε, τα βίντεο δεν τα έχουμε γράψει στο δισκάκι, μπορείτε να τα βρείτε στο, στο πόρταλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή. Μπορέσαμε να μάθουμε τι ισχύει σε αυτή την ε, απότερη περιφέρεια, τα συγκεκριμένα προβλήματα, πάρα πολύ θετικά αυτά. Περάσαμε καλά πέραν των άλλων, παρά το ότι δουλεύαμε μέρα και νύχτα. Όλοι, όλοι, όπως είπατε, βουλευτές, διερμηνείς, όλοι. Ε, δημιούργησε ένα κλίμα πάρα πολύ ευχάριστο. Βεβαίως και ευχαριστούμε για τα όσα μας εξηγήσατε αλλά πρέπει και τους διερμηνείς να ευχαριστήσω. Γιατί όπως πάντα μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και οι επικεφαλής της γραμματείας. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για αυτή την σύνοψη της ε, δραστηριότητας αποστολής. Βοήθησαν λοιπόν όλοι πάρα πολύ. Και επομένως η κατάληξη ήταν πάρα πολύ θετική. Σας ευχαριστώ όλους. Οι συζητήσεις ήταν πάρα πολύ ζωηρές. Και βέβαια, και εγώ ως Ισπανίδα, είχα πολλά να συζητήσω. Γιατί και εμεί έχουμε κοινά προβλήματα, έχουμε και εμεί από την περιφέρεια, τα Κανάρια. Πάρα πολύ θετική αυτή η αποστολή. Ευχαριστώ πάλι. Το τελευταίο τώρα σημείο. Γιατί έτσι, αν το συζητήσουμε, θα έχουμε ένα μεγάλο διάλειμμα και θα ξαναπούμε τα πούμε στις 3 ε, η ώρα με την έκθεση του κυρίου Βαλέσα. Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε στις 3 η ώρα.